morning, Καλώς ορίζατε στο δεύτερο τμήμα της τακτικής συνεδρίασής μας της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Σήμερα το πρωί θα ξεκινήσουμε με το σημείο 12. Θα εξετάσουμε την ερώτηση με την προφορική απάντηση σε σχέση με την ανατολική εταιρική σχέση. Φυσικά πρόκειται για εμπορικά θέματα. Πριν από την ε, Σύνοδο στο Βίλνιους, αργότερα φέτος, η κυρία Ερικενέ είναι η συγγήτρια και θα της δώσω το λόγο. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, όπως ε, ξέρετε, η Σύνοδος Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης θα λάβει χώρα στη ε, Λιθουανία στα τέλη Νοεμβρίου και θα καθορίσει αν η ανατολική εταιρική σχέση μπορεί να θεωρηθεί ως επιτυχία, κυρίως ε, σε ό,τι αφορά της, ε, το να ενταχθούν οι χώρες της ε, περιοχής στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω σφαιρικών και συμβάθων συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών. Αυτή η προφορική ερήτηση που ελπίζω να εθετήσουμε σήμερα σε αυτή την Επιτροπή ελπίζω να οδηγήσω στο να έχουμε αυτή την προφορική ερώτηση στο Στρασβούργο στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Με αυτή την ερώτηση θα ζητήσω από την Κομισιόν να μας παρουσιάσει ποιες είναι οι προοπτικές και ποια βήματα θα ληφθούν κατόπιν της Συνόδου Κορφή. Κάθε εμπορική σχέση είναι πολύ διαφορετική και επομένω η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μπορεί να έχει μια ξεκάθαρη μακροπρόθεσμη στρατηγική για την εμπορική και οικονομική σύνδεση με τις χώρες αυτές. Από καταλαβαίνω, αν και αυτές οι χώρες βρίσκονται σε εντελώς διαφορετικά στάδια της διαδικασίας ολοκλήρωσης και έχουν εντελώς διαφορετικές οικονομικές ανάγκες και εμπορικά συμφέροντα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν και διαφορετικές προσδοκίες για τις εμπορικές τους σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Λευκορωσία και το Αζερβαϊτζάν ξεχωρίζουν γιατί ποτέ δεν έχουν μπει στη διαδικασία σύνδεση. Η Λευκορωσία δεν είναι ενεργή στην ανατολική εταιρική σχέση, ενώ το Αζερβαϊτζάν δεν ανήκει στον ΠΟΕ και δεν έχει πρόθεση να συμμετάσχει βραχυπρόθεσμα. Επομένω, δεν μπορεί να διαπραγματευτεί μια σφαιρική και σεβατό συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, επικεντρωνόμενη στι ε, ε, συμφωνίε με ε, τη Γεωργία, τη Μολδαβία, την Ουκρανία. Η ερώτηση αφορά τα εξή. Καταρχήν το θέμα τη υπογραφή και τη εφαρμογή αυτών των ε, συμφωνιών ελευθερών συναλλαγών και κατόπιν το πρόβλημα τη παρέμβαση τη Ρωσία και των επιλογών των χωρών αυτών. Ουκρανία. Καθώ η DCFTA με την Ουκρανία μονογράφηκε ήδη πριν 14 μήνε, η υπογραφή τη συμφωνία βρίσκεται στην ατζέντα της Συνοδού αν θα δεχτούει τελικά ε, η Ουκρανία να εφαρμόσει τις συνθήκες που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν και κάποιες ανησυχίες ε, προστατευτισμού στην Ουκρανία που μάλλον δεν θα εξαφανιστούν εν μία νυχτή ακόμη και αν υπογραφεί η Συμφωνία Σύνδεσης. Επομένως, η ερώτησή μου το χάρη είναι πώς η Κομισιόν μπορεί να ξεκινήσει την εφαρμογή της DCFTA σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Ουκρανίας και πώς ε, παραδείγματος χάρη ε, θα πείσει να εγκαταλειφθούν ε, κάποιες πολιτικές παραδείγματος χάρη όπως το τέλος ανακύκλωσης επί των οχημάτων. Επίσης ανησυχώ για τις συμφωνίες με Αρμενία, Γεωργία και Μολδαβία. Οι διαπραγματεύσει ολοκληρώθηκαν πριν από τι καλοκαιρινέ διακοπέ με τι χώρε αυτέ. Νωρίτερα αυτό μήνα, ο πρόεδρο τη Αρμενία ανακοίνωσε ότι θα μπει η χώρα του στην Ευρωασιατική Τελωνική Ένωση και η Κομισιόν δεν έχει αντιδράσει ακόμη και δεν έχει εξηγήσει πώ θα προχωρήσει με τη διαπραγμάτευση αυτή τη συμφωνία για τη Γεωργία και τη Μολδαβία υπάρχουν παρόμοιες πιέσεις από τη Ρωσία στις ε, χώρες αυτές ε, και αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν ε, κάποιες επικράτειες όπου δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί η συμφωνία. Πρέπει να προωθηθούν τα πλεονεκτήματα της συμφωνίας σε σχέση με το να συμμετέχουν στην Τελωνιακή Ένωση οι χώρες αυτές και θα πρέπει να εφαρμοστεί η συμφωνία παρά τις πιέσεις και τις διαφωνίες. Οι DCFTAs αποτελούν τον ακρογωνίο λίθο της ε, ε, Ανατολική Εταιρική σχέση ε, και υπάρχει ένα κίνδυνο να μην έχει τα απαιτούμενα αποτελέσματα η Συνοδός αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιταχύνει τη διαδικασία και λάβει συγκεκριμένα βήματα. Διαπραγμάτευση μια συμφωνία είναι το ένα, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επίση να διασφαλίσει ότι είναι πεπισμένη η εταίρεια ότι η CFTA είναι απαραίτητο βήμα προ την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση που θα ωφελήσει την οικονομία και του πολίτε και για του λόγου αυτού αυτέ οι συμφωνίε θα πρέπει να εφαρμοστούν πλήρω με την αρρωγή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτή την προφορική ερώτηση πιστεύω ότι αυτή η Επιτροπή μπορεί να ασκήσει πίεση στην Κομισιό να λάβει περισσότερε πρωτοβουλίε προ αυτήν την κατεύθυνση και τώρα αλλά και μετά τη Σύνοδο Κορφή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ας αρχίσουμε τη συζήτηση. Η ερώτηση υπάρχει στο φάκελό σα. και ας αρχίσουμε τους του συζητητές. Α, δεν... Ε, Ας αρχίσουμε λοιπόν τους σκιώδεις εισηγητές. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και την ομιλήτρια για την ενδελεχή αναφορά και σκιαγράφηση της κατάστασης. Πιστεύω ότι αυτή η προφορική ερώτηση είναι, έρχεται την κατάλληλη στιγμή για να ζητήσουμε μία απάντηση, μία αντίδραση σε αυτό το ζήτημα. Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι είναι πολύ σημαντική η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο να μην ξεχνάνε την κατάσταση που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή με τη Ρωσία, διότι προφανώς η Ρωσία επιζητεί τη δημιουργία μιας νέας τελωνιακής ένωσης και ε, πρώην, χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης έχουν ορισμένες ε, αδυναμίες παρόλο τις στενές σχέσεις που έχουν με τη Ρωσία. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει εμείς να κοιτάξουμε να βρούμε την πιο αποτελεσματική οδό για να πείσουμε αυτή τη χώρα να εξακολουθήσει να μένει στην Ευρωπαϊκή Οδό, να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Οδό και κατεύθυνση. Επίσης, από την άλλη πλευρά, είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχάσουμε τις καλές σχέσεις με τη Ρωσία, ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για μας. Νομίζω ότι η Ρωσία χρειάζεται την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρώπη και αντίστοιχα και παίζοντας ε, αυτό το παιχνίδι στις σχέσεις μας ε, πρέπει να δούμε πώς θα διαμορφώσουμε την διαπραγματευτική μας ε, γραμμή και να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες μαζί με τη Ρωσία. Ας δούμε πώς θα απαντήσει, πώς θα αντιδράσει η Κομισιόν σε αυτή την προφορική ερώτηση. Ο πρόεδρος, η, η ο Γιάννη Κλαντό από τους Πράσινους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον, την εισηγήτρια, η οποία νομίζω εξήγησε αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους πρέπει να υποβληθεί αυτή η προφορική ερώτηση. Από την πλευρά των πρασίνων, δεν θεωρούμε ότι είναι και κέρια η σκόπιμη αυτή η ερώτηση αυτή τη στιγμή. Στην τελευταία ολομέλεια υπερψηφίστηκε ε, ένα ψήφισμα για την ε, ανατολική συνεργασία με το οποίο καταδικάζαμε την πίεση από τη Ρουσία και εδώ θα βρισκόμαστε σε μια συζήτηση σχετικά με την Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου ενώ στην πραγματικότητα το ερώτημα, το ζήτημα είναι πολιτικό. Δεν βλέπω λοιπόν πως μέχρι να βελτιωθεί η πολιτική κατάσταση, οι πολιτικές σχέσεις, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε ενίσχυση της ε, ε, Συζήτηση ε, των διεργασιών για τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου. Αυτή είναι η θέση των πρασίνων, δηλαδή εμεί πιστεύουμε ότι το ζήτημα δεν είναι τόσο, μάλλον είναι περισσότερο, να δούμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει την Ουκρανία έναντι της Ρωσίας, αλλά επίσης πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει την Ουκρανία στην υλοποίηση των κριτηρίων που συμφωνήθηκαν το 2012. Επομένως, από την πλευρά τους οι πράσινοι δεν υποστηρίζουν ε, και τόσο αυτήν την προφορική ερώτηση. Θεωρούμε ότι είναι άσκοπη και δεν έρχεται σε κατάλληλη χρονική στιγμή. Ευχαριστούμε. Η Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς ο σκιώδης ηγητής μας δεν είναι εδώ που ασχολείται κυρίως με την οικονομική πτυχή. για. αυτό αυτό θέλω και μετά από τη συζήτηση στην Ολομέλεια που έγινε την περασμένη εβδομάδα να συμπληρώσω κάτι. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για την εκτενή εργασία την οποία έκανε και την εξαιρετική εισαγωγή στο θέμα και περιγραφή του θέματος. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με τους, ε, ε, με τις χώρες που έχουμε εταιρική σχέση, τις ανατολικέ χώρες. Όποιος παρακολούθησε τη συζήτηση την περασμένη Τετάρτη πιστεύω ότι είδε σαφώς ότι δεν έχουμε ακόμα καταλήξει, δεν έχουμε φτάσει στην βέλτιστη κατάσταση. Δεδομένου ότι όταν μιλάμε για οικονομικά θέματα πάντοτε θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τη σχέση μας με τη Ρωσία το θέμα ότι βεβαίως κάθε χώρα ε, της ανατολικής εταιρικής ε, σχέσης έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει τη δική της πολιτική, τις εξωτερικές σχέσεις, τις εμπορικές ε, διαπραγματεύσεις κλπ. Σωστό, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να περιμένουμε τη σύνοδο κορυφή στο Βίλνιος μέχρι ότου εμείς ως Επιτροπή ΙΝΤΑ έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα όλης της κατάστασης, όλου του θέματος. Οπότε τότε θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε την Κομισιόν με τα συμπεράσματα του Βίλνιους, διότι ξέρουμε ότι στο Συμβούλιο υπάρχουν μεγάλες διαφορές απόψεων, δηλαδή το θέμα του πώς θα αντιμετωπίσει το Συμβούλιο και τι θα αποφασίσει για τη μελλοντική διαμόρφωση των εταιρικών σχέσεων με τις ανατολικές αυτές χώρες δεν έχει τελειώσει, δεν έχει ολοκληρωθεί. Γι' αυτό πρέπει μετά να προσεγγίσουμε και να ξανααποτανθούμε ε, στην Κομισιόν, μετά το Βίλνιος. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ε, τέλος, ο Μπέρτ Λάγκε, τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ θερμά την εισηγήτρια για το σχέδιο αυτό της ερώτησης, πιστεύω ότι ο Χέλμουτ ε, έθεσε τον δάκλειο των τύπων των δήλων. Διότι πρέπει να περιμένουμε στο Βίλ... τι θα γίνει στο Βίλνιους και να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να ληφθεί μια θετική απόφαση. Να μην ε, οικοδομούμε, να μην φτιάχνουμε καταστάσεις οι οποίες μετά δεν στέκονται σε εθνικό επίπεδο. Ε, μην ξεχνάτε και την υπόθεση Τιμοσέγκο, παρόλο που πρέπει να συζητήσουμε την... Ε, ε, ξέρουμε ότι δεν είναι και άγια η γυναίκα, εν πάση περιπτώσει, δεν πρέπει να θέτουμε εμείς προσκόμματα στις δικές μας εργασίες, στα δικά μας θέματα επισημούμε μια στενότερη συνεργασία με την Ουκρανία. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτή είναι η ουσία, δεν είναι. Είναι, είναι ε, το 85% του ΑΕΠ όλης αυτής της περιοχής προέρχονται από την Ουκρανία. Είναι δηλαδή η πιο σημαντική χώρα αυτής της περιοχής του κόσμου. Και γι' αυτό βεβαίως θέλουμε επί τη βάση των δικών μας αρχών να δημιουργήσουμε στενότερη εμπορική σχέση. Ε, πρέπει όμως να δούμε και τι θα γίνει στο Βίλνιος έτσι ώστε να μπορούν και εμπορικές διαπραγματεύσεις να είναι βιώσιμες, υλοποιήσιμες. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Να ακούσουμε τώρα την Επιτροπή, τη γνώμη της Κομισιόν. Διότι αυτό είναι ένα ζήτημα που απευθύνει στην Κομισιόν. Ο κύριος Ντεβίνιε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για τις λίγαν επίκαιρες ε, ερωτήσεις, τα, τα επίκαιρα αυτά θέματα ε, που αφορούν τη σημερινή κατάσταση. Ε, θα, θα απαντήσω στις ερωτήσεις. Όσον αφορά την Ουκρανία, ξέρετε ότι έχουμε μια ιδιαίτερη κατάσταση όσον αφορά τα πολιτικά κριτήρια τα οποία έθεσε το Συμβούλιο. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να αντιμετωπίσουμε την υπάρχουσα συμφωνία η οποία υπάρχει με την Ουκρανία σήμερα. Αυτά τα δύο δεν αντιμάχονται, δεν είναι αντίθετα, διότι αυτή τη στιγμή ακολουθούμε την ε, ατζέντα για τα DSFTAs, ε, και πιστεύω ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις θα διευκολύνουν την επίλυση ορισμένων διαφορών που εκκρεμούν. Πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε αυτή την παράλληλη πορεία. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε αιτήματα των χωρών αυτών για επιτάχυνση της διαδικασίας και για υπογραφή των DSFTAs, των ε, ε, συμφωνιών για τις ζώνες των αλλαγών και όπως ξέρετε οι διαδικασίες μας και στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν συνεχίζονται και κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο. Τέλος, όσον αφορά τις σχέσεις με τη Ρωσία που αναφέρθηκαν πολλαπλώς, καταρχάς, ας μην ξεχνάμε ότι ό,τι πράττουμε με τους ανατολικούς εταίρους δεν θα πρέπει να έχει καμία αρνητική επίπτωση, αντίκτυπο ως προς τη Ρωσία. Και αυτό ισχύει, διότι κανένα από τα DCFTAs και τις διαπραγματεύσει που, και που κάνουμε ή που έχουμε με τους ανατολικούς εταίρους ε, έχουν αρνητικές επιπτώσεις ή αντίκτυπο στη Ρωσία. Τώρα βέβαια το να δημιουργηθεί μια νέα τελωνιακή ένωση και να είναι κάποιος, να γίνει κάποιος μέλος σε μια νέα τελωνιακή ένωση με τη Ρωσία είναι εντελώς άλλο ζήτημα, διότι αυτό εμποδίζει την υπογραφή του DCFTA. Δεν έχουμε καμία πρόθεση βεβαίως να ε, προχωρήσουμε εναντίον της Ρωσίας ή να προσφύγουμε κατά της ε, Ρωσίας. Το αντίθετο, διότι χαιρόμαστε ιδιαίτερα που εξυγχρονίζεται η οικονομία της και οι προσπάθειες που κάνει. Αλλά έχουμε δει ότι υπάρχει η η Ρωσία ασκεί μεγάλες πιέσεις έναντι αυτό το χρόνο και αυτές οι πιέσεις που ασκούνται τελευταίως είναι απαράδεκτες και γι' αυτό ακριβώς θέλουμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Ο πρόεδρος δεν απαντήσετε για την Αρμανία που επί της οποίας σιωπή η Κομισιόν μετά τη δήλωση της Ρωσίας ότι αποφάσισε να συνυπογράψει την Τελωνιακή Ένωση για την Αρμενία η Κομισιόν. Πιστεύω ε, η Κομισιόν έκανε μια δήλωση, εμείς παρακολουθούμε την κατάσταση της εξελίξης στην Αρμενία, ε, είναι στη διάθεσή τους να ακολουθήσουν τι πολιτική, οικονομική και εμπορική επισημούν. Από σας είπα, ορισμένες επιλογές ε, δεν συνάδουν με την Τελωνιακή Ένωση ή με την ατζέντα των DCFTA. Δυστυχώς αυτή είναι η περίπτωση με την Αρμενία. Εάν προσχωρήσει στην Τελωνιακή Ένωση θα πρέπει να αυξήσει τους δασμούς. Δυστυχώς, αντί αν υπογράψει το DCFTA θα έχει τη δυνατότητα να μειώσει τους δασμούς, να, να εφαρμόσει ορισμένα ε, πρότυπα ε, για την ασφάλεια υγείας και τροφίμων και πολλά άλλα πλεονεκτήματα τα οποία θα ενισχύσουν την ασφάλεια των τροφίμων και άλλα συναφή θέματα. Γι' αυτό ακριβώς επισημούμε εμείς να ακολουθήσει το, το, τις διαπραγματεύσεις του DCFTA και να συνυπογράψει. Ε, αλλά βεβαίως δεν μπορούμε να επηρεάσουμε από εμπορική άποψη, απόψεως τις επιλογές της Αρμενίας. Ωραία. Να επανέλθουμε στην εισηγήτρια. Κυρία Αντρικένε, για τελικά σχόλια έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Κιωδείς και τους συντονιστές από όλες τις πολιτικές ομάδες ε, για τις απόψεις που εξέφρασαν. Και θα ήθελα και να τονίσω ότι έχουμε σχεδιάσει αυτή την προφορική ερώτηση εδώ και καιρό. Αρχίσαμε να εργαζόμαστε από αυτού πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές και τώρα που πλησιάζει η Σύνοδος Κορφής πρέπει να ακούσουμε τον Επιτροπό Δεγκούχτ για τις σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και τις δράσεις που αναλυθούν πριν και μετά τη Σύνοδο σε ό,τι αφορά το ψήφισμα που υιοθέτησε την περασμένη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νομίζω ότι περισσότερο ήταν πολιτική δήλωση και δεν επικεντρωνόταν στις ε, DCFTAs, αλλά καθώς εμείς είμαστε η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, πρέπει και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Και συνάδελφοι που ενδιαφέρονται από άλλες επιτροπές ε, θεωρούν ε, και εγώ θεωρώ ότι θα ήταν ε, πολύ καλό να προχωρήσουμε τον Οκτώβριο. Κύριε Σόλτς, έχετε ζητήσει το λόγο. Ναι, μετά το σχόλιο της Κομισιόν αναρωτιέμαι και με συγχωρείτε γιατί έχω μια ακόμη ερώτηση για το θέμα. Αν κατάλαβα πλήρως την περιγραφή σας της Τελωνιακής Ένωσης αλλά από την νομική σκοπιά, για αυτή την τηλεονική ένωση που του είναι διαπραγματεύσεις, ε, πώς ε, θα είναι και οι σχέσεις με την Τουρκία και γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις ακολουθούμε μια συγκεκριμένη διαπραγματευτική διαγραμμή και σε άλλες περιπτώσεις άλλη. Κομισιόν, μπορείτε να αντιδράσετε σύντομα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κατάσταση διαφέρει με την Τουρκία. Γιατί η Τουρκία είναι σε τελωνική ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι ασύμμετρη. Δηλαδή η Τουρκία έχει δεσμευτεί να αναλάβει τις προτιμήσεις που διαπραγματεύεται την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχει το αντίστροφο. Πρόκειται λοιπόν για μια διαφορετική κατάσταση από μια κλασική τελωνική ένωση που έχουμε εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω ξέρετε, η εμπορική πολιτική ασκείται ολοκληρωτικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ψηφίσουμε Αργότερα αυτή την προφορική ερώτηση βρίσκεται στον κατάλογο ψηφοφοριών. Περνάμε στο σημείο 13. Και πάλι επανερχόμαστε σε αυτό το σημαντικό φάκελο σε ό,τι αφορά την ε, αμοιβαιότητα στις δημόσιες συμβάσεις και την πρόσβαση εταιριών τρίτων χωρών στις δημοσίες συμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ξέρετε, αυτό το θέμα το συζητάμε εδώ και ένα χρόνο σχεδόν και έχουμε ανταλλάξει απόψεις πολλάκις. Ο εισηγητής έχει παρουσιάσει το το οποίο έχει συζητηθεί. Και τώρα έχουμε το σχέδιο της έκθεσης. Και φυσικά πρέπει να τη συζητήσουμε. Ο κύριος ε, Κασπάρη είναι εισηγητής, ζητά συγγνώμη όμως που δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Ξέρετε γιατί, λόγω προεκλογικής εκστρατείας στη Γερμανία. Παρ' όλα αυτά θα αντικατασταθεί από κάποιο συνάδελφο που θα μας παρουσιάσει το ε, σχέδιο έκθεσης του κυρίου Κασπάρη και φυσικά θα του γνωστοποιήσει και το τι θα προκύψει από τη συζήτησή μα. Έχω συμφωνήσει για τη στρατηγική, ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό ο φάκελο και μα πιέζει ο χρόνο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Αξιότιμε πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, Ασφαλώς όλοι βρισκόμαστε σε υποκλοϊκό περίοδο στην ε, Γερμανία και ο Ντανιέλ Κασπάρη, αλλά σήμερα δυστυχώς ο συνάδελφός είναι στο, έπρεπε να είναι στο νοσοκομείο και δεν μπόρεσε να αναβάλει αυτή την, ε, ε, ε, κάνει μια χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο και δεν μπορούσε να την αναβάλει. Γι' αυτό μου ζήτησε να παρουσιάσω πολύ σύντομα το θέμα του, το, το οποίο νομίζω επί της ουσίας το γνωρίζουμε. Είναι μια τελείωτη συζήτηση αυτή και ο εισηγητής λέει σαφέστατα ότι μετά από την τελευταία ανταλλαγή απόψεων στο Συμβούλιο δεν έχει επέλθει καμία τροποποίηση. Δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά σε, αυτούς, σε αυτά τα σχέδια κανονισμού συμβαίνει αυτά συχνά. Υπάρχουν κράτη-μέλη που υποστηρίζουν την πρόταση της Κομισιόν. Μία εισάρισμη μερίδα, ένα ομάδα κρατών μελών δεν υποστηρίζει την πρόταση διότι πιστεύουν ότι είναι υπερβολικά προστατευτική αυτή η πρόταση. Έχει δηλαδή στοιχεία προστατευτισμού και γι' αυτό θα έχει αρνητικά αντίκτυπο στο διεθνές εμπόριο και ενδεχομένως αντίπεινα. Και η τρίτη ομάδα πιστεύει ότι κάτι μπορεί να γίνει, αλλά όχι με αυτή τη μορφή που προτείνεται. Έχουμε λοιπόν την κλασική περίπτωση τριών διαφορετικών απόψεων. Το ίδιο ισχύει και για την Επιτροπή μας. Ορισμένοι θέλουν να γίνει πιο, αυστηρό, πιο αυστηρή η πρόταση, α, σε άλλους δεν αρέσει καθόλου και η τρίτη ομάδα λίγο πολύ συμφωνεί στις βασικές αρχές. Αυτό το οποίο πιστεύω ότι όλοι θέλουν είναι να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε μέσω αυτού του κανονισμού να μην δημιουργηθεί καμία στρέβλωση ή αντιφάσεις στην εσωτερική αγορά της Ένωσης. Εδώ λοιπόν έχει ο εισηγητής προσπαθήσει να συγκεράσει τις διαφορετικές απόψεις. Έχετε την έξεση. ελπίζω, τουλάχιστον εγώ την έχω. Και ε, στο πρώτο έγγραφο εργασίας ο εισηγητής έθεσε 5-6 ερωτήσεις και ζήτησε ε, από τους συναδέλφους να μελετήσουν αυτά τα θέματα που έθεσε με τις ερωτήσεις για να μπορέσει να συντάξει την έκθεσή του. Ο, σε, ο, ο, κύριος, ο συνάδελφος μας, κύριος Κασπάρης, θέλει να τονίσει ορισμένες πτυχές. Πιστεύω ότι η πρόταση της Κομισιόν δεν απαντά στο ερώτημα εάν θέλουμε άνοιγμα των, δημοσίων, των αγορών δημοσίων συμβάσεων, αν θέλουμε αυτό το άνοιγμα ή εάν δημιουργείται μέσω των, προ, των προτάσεων του κανονισμού ένα μέσο προστατευτισμού. Κατά την αντίληψή μου υπάρχουν επιχειρήματα που υποστηρίζουν και τις δύο κατευθύνσεις. Αλλά η Κομισιόν δεν αναφέρεται στους στόχους ε, αυτού του κανονισμού. Ε, δεν είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό ο εισηγητής έχει επιφυλάξει στο να απορρίψουμε το σύνολο του κανονισμού και γι' αυτό επισημεί την εισαγωγή μιας ρήτρας αναθεώρησης έτσι ώστε η Κομισιόν μετά από μια συγκεκριμένη προθεσμία να μπορεί να επανεξετάσει, να αναθεωρήσει και να αξιολογήσει τι έχει συμβεί και εάν πράγματα, πράγματι έχουν ανοίξει οι αγορές δημοσίων συμβάσεων ή έχουν περιοριστεί περισσότερο με προστατευτικά μέσα. Ο κύριος Κασπάρη επίσης προτείνει η θέση ενισχύ της εκτελεστικής πράξης να διαρκεί τουλάχιστον ε, το, το πολύ πέντε χρόνια. Πέντε χρόνια η διάρκεια της εκτελεστικής πράξης ε, δεδομένου ότι υπάρχει περίπτωση να θέτει ορισμένα περιοριστικά μέτρα και να επιβάλλει ορισμένα μέτρα περιοριστικής μορφής. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει να ισχύει για πάνω από πέντε χρόνια ε, η εκτελεστική πράξη. Ωραία και καλά όλα αυτά, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε το στόχο. Και μετά βάσει του στόχου που έχουμε μπορούμε να κοιτάξουμε πώς θα προχωρήσουμε. Τώρα, το θέμα των αναπτυσσομένων χωρών. Βεβαίως υπάρχει ο κίνδυνος, οι αναπτυσσόμενες χώρες να γίνουν θύματα αυτού του μέσου. Και εδώ πάλι δεν, ε, δεν καινοτομούμε, δεν είναι κάτι το καινούργιο αυτό, διότι ξέρουμε ότι υπάρχουν αναπτυσσόμενες χώρες που δεν είναι σε θέση να ανοίξουν την αγορά δημοσίων συμβάσεων και ορισμένες φορές οι λιγότερο επιτυγμένες χώρες ούτε καν διαθέτουν αγορά δημοσίων συμβάσεων. Το θέμα είναι οι λιγότερες ανεπτυγμένες χώρες να μην καλυφθούν από το πεδίο ισχύω και να εξαιρεθούν και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες. Δηλαδή προτείνει ο εισηγητής να εξαιρεθούν ορισμένες λιγότερο ανεπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες χώρες, βεβαίως ε, πάντοτε σύμφωνα με την ε, εμπορική μας πολιτική και θα πρέπει οι, τα θεμελιώδεις αρχές της ευρωπαϊκής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάντοτε να εφαρμόζεται και πάντοτε να συνάδει με τις συμφωνίες που γίνονται με αυτές τις χώρες. Ε, να μην παρεκκλίνουμε δηλαδή ε, από την εμπορική μας πολιτική και να είμαστε πάντοτε συνεπείς προς αυτήν. Το τρίτο θέμα, η ομοιομορφία της ε, κοινή ε, εμπορικής πολιτικής. Δεν θα πρέπει ε, με κανένα τρόπο να υπονομευθεί αυτή η ομοιομορφία της, του χειρισμού. Ξέρουμε ότι σε ορισμένε χώρες υπάρχουν εθνικές ρυθμίσεις, εθνικές διατάξεις που μπορούν να δημιουργήσουν ε, μία στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς. Ε, δεν είναι δυνατόν ε, ορισμένες συμφωνίες δημοσίων συμβάσεων να στρεβλώσουν την εσωτερική αγορά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το λέει σαφέστατα ο κανονισμός ότι τα κράτη-μέλη δηλαδή οι οι αναθέτουσες αρχές των κρατών μελών θα επιτρέπουν την πρόσβαση προϊόντων και υπηρεσιών από τρίτες χώρες μόνον όταν υπάρχει ο κίνδυνος στρέβλωσης ή κατακαιρματισμού της εσωτερικής αγοράς. Και η πρόταση του εισηγητή είναι η εξής. Λέει ότι η πρόταση της Κομισιόν, όπως είπαμε, μπορεί να οδηγήσει σε μία διάσπαση, σε έναν κατακαιρματισμό της εσωτερικής αγοράς όταν ένας ε, πλειοδότης κάνει μία προσφορά η οποία δεν μπορεί, αποκλείεται από την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι παραδεκτή, αλλά ταυτόχρονα έχει κάνει ο πλειοδότης και μία άλλη προσφορά σε, μια, σε ένα άλλο κράτος μέλος. Από το ένα λοιπόν κράτος απορρίπτεται, ενώ στο άλλο επιτρέπεται να υποβάλει την προσφορά του. Αυτό θα οδηγήσει σε στρεβλώσεις της εσωτερικής αγοράς και γι' αυτό η αναθέτους λέει ο συγητής ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση του πλειοδότη ε, σε δημόσιες συμβάσεις όταν η Κομισιόν έχει κάνει μία εξέταση του θέματος και έχει διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει αμοιβαιότητα στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ της χώρας του πλειοδότη και της χώρας της αναθέτουσας αρχής. Άμα δεν υπάρχει αυτή η αμοιβαιότητα δεν προχωρούν οι δημόσιες συμβάσεις, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μέσω της Επιτροπής μία συνεχής και προσεκτική παρακολούθηση, εποπτεία ε, της αυτή αυτής και της συμπεριφοράς των ε, κρατών των πλειοδοτών. Ε, έχει λοιπόν μία ε, μεγαλύτερη ευθύνη η Κομισιόν ως προς αυτό το ζήτημα. Εάν λοιπόν δεν δικαιολογείται ή ε, ο περιορισμός, η περιοριστική εφαρμογή του κανονισμού αυτού, αυτού δεν μπορεί να εφαρμοστεί από την αναθέτουσα αρχή. Εάν όμως υπάρχουν βάσιμοι, βάσιμοι λόγοι μπορεί να περιοριστεί η περιοριστικη εφαρμογη του κανονισμου αυτου δεν μπορει να εφαρμοστει απο την αναθετουσα αρχη εαν ομως υπαρχουν βασιμοι λογοι μπορει να περιοριστει η προσβαση Εάν παρακολουθώντα τώρα την αγορά δημοσίων συμβάσεων, τουλάχιστον στη δική μου περιφέρεια, δεν νομίζω ότι καθένα έχει διάθεση ή ε, όρεξη να υποβάλει οποιαδήποτε ε, να υποβληθεί σε οποιοδήποτε έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιοριστικές αποφάσεις. Δεν νομίζω ότι θα, θα, θα έχει το, τη διάθεση να συμμετάσχει σε ένα δημόσιο, σε μια πλειοδοτικό διαγωνισμό σε δημόσια σύμβαση αν γνωρίζει ότι θα υποβληθούν περιοριστικοί όροι. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο Ντανιέλ Κασπάρη έχει υποβάλει μια πολύ σωστή και <clears throat> προσεκτικά μελετημένη πρόταση έχοντας συγκεράσει όλες τις ε, απόψεις και τις διαφορετικές ε, πτυχές και τον, θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά για την εργασία του αυτή. Σας ευχαριστούμε για αυτή την ξεκάθαρη και εκδοτική παρουσίαση της εκθέσης του κ. Κασπάρη. να σας πω ότι δεν ήξερα ότι ο κ. Κασπαρία έλειπε για λόγους υγείας και ελπίζω να του διαβιβάσετε τις ευχές μου για περαστικά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Κύριε και ο κ. Λάγκε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την συνάδελφό μας για την παρουσίαση του, της προτάσεως αυτής. Οχτώ σημεία μου έχουν, πιστεύω ότι αξίζει να συζητηθούν ή τα οποία ε, αξίζουν της υποστήριξή μας. Καταρχάς ο κύριος Κασπάρη προτείνει το πεδίο εφαρμογής σε τρίτες χώρες που είναι ιδιαίτερα δύναμες να εξαιρεθούν. Να υπάρχει λοιπόν εξαίρεση των λιγότερων ανεπτυγμένων από τι ανεπτυσσόμενες χώρες. Εξαίρεση, ρήτρα εξαίρεση. Δεύτερον, η σχέση μεταξύ του άρθρου 6 και του των άρθρων 8 και 10. Δηλαδή, όταν περιφερειακές αρχές αποκλείουν πρόσβαση την πρόσβαση, πώς εμπλέκεται η Κομισιόν. Ο κύριος Κασπάρη προτείνει όταν η Κομισιόν κάνει μια μελέτη, μια έρευνα των προσφορών και δει ότι τα πράγματα δεν είναι σωστά, τότε μπορεί η αναθέτουσα αρχή να αποκλείσει την πρόσβαση. Εγώ το βλέπω αντίθετα. Όταν αναθέτουσες αρχές αποκλείουν πλειοδότε, τότε, τότε θα πρέπει η Κομισιόν να ξεκινήσει την έρευνα. Γιατί και πώς. Αυτό μου φαίνεται εμένα πιο λογικό για να δούμε ακριβώς ε, τι σχέση υπάρχει μεταξύ της υποβολής και του αποκλεισμού. Δεδομένου ότι υπάρχουν ε, τοπικές αρχές, τοπική αυτοδιοίκηση ας πούμε, που είναι αναθέτους αρχή, που δεν μπορεί να είναι εν γνώση όλων των ε, περιπλοκότητων που υπάρχουν στις διαδικασίες κομισιών. Τρίτον, ο εποπτική, εποπτικός ρόλος της Κομισιόν, αυτό το υποστηρίζουμε. Πρέπει να υπάρχει αυτή η εποπτεία και, να είναι και γρήγορα, ταχεία. Τέταρτον, αυτή η νομοθεσία, αυτό το μέσον, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την αηφορία, ιδιαίτερα στο θέμα των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των κοινωνικών συνθήκων εργασίας. Και προτείνουμε η... το αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου μεταξύ Κοινοβουλίου Συμβουλίου όσον αφορά το θέμα των αναθέσεων ιδίως στο άρθρο 41 ε, και 15, να χρησιμοποιηθούν, να ενσωματωθούν εδώ ως κριτήρια και τα άρθρα αυτά να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν την αξιολόγηση των, ε, της, της χρήσης των ε, θεμελιωδών αρχών. Δηλαδή να αξιολογήσουν αν έχουν πραγματικά ληφθεί υπόψη οι θεμελιώδεις αρχές εργασίας και κοινωνικών προτύπων. Πέμπτον, ο εισηγητής λέει ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα αναθεώρησης ε, του κανονισμού το πολύ ε, μέσα σε πέντε χρόνια ε, με προθεσμία πέντε ετών. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να περιορίσουμε ούτε τη χρονική διάρκεια ούτε το εύρος της αναθεώρησης πρέπει να αξιολογήσουμε ε, και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Ενδέχεται στο τέλος να καταλήξουμε ότι τα μειονεκτήματα είναι περισσότερα από τα ωφέλη αυτής της, ε, του κανονισμού και μήπως θα πρέπει να προχωρήσουμε μετά σε άλλη κατεύθυνση. Έκτον, τροπολογία 25. Ε, all που λέει ότι όλες οι χώρες με τις οποίες διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξαιρεθούν. Η Κομισιόν λέει ότι μόνο όταν πρόκειται για ουσιαστικές ε, διαπραγματεύσεις. Εμείς ξέρουμε ότι ήδη γίνονται διαπραγματεύσεις με πολλές χώρες και πιστεύω ότι αυτή η πρόταση για ουσιαστικές πραγματεύσεις είναι παράλογη. Τέλος, όταν αποφασίζουμε ε, νομοθετικές ε, πράξεις πρέπει να δούμε ε, πώς θα υπάρξει μια δημόσια σύμβαση μεταξύ μιας χώρας ας πούμε και μιας πόλης, της Βαρκελόνης και πώς αν κάποιος υποβάλλει ε, μια πρόταση στη Βαρκελόνη δεν την υποβάλλει και κάπου αλλού. Εκεί έχει δίκιο ο κύριος Κάσπαρη να μην υπάρχει αυτός ο κατακαιρματισμός και η στρέβλωση. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, την προστιθέμενη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό αυτό το ομοχρό της προστιθέμενης αξίας πρέπει επίσης να ενσωματωθεί σε αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. Όχι, δεν είναι εδώ από τους φιλελευθέρους, από το ECR, Ευρωπαίοι Μεταρρυθμιστικές Συντηρητικέ. παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, βρισκόμαστε άλλη μια φορά να συζητάμε αυτό το αμφιλεγόμενο θέμα. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή που ασχολείται με αυτό το δύσκολο ζήτημα. Και παρά το γεγονό ότι εγώ διαφωνώ από... με διάφορες ε, θέσεις που έχουν εκφραστεί σε αυτό το θέμα, συνεχίζω να ασχολούμαι με αυτό το φάκελο. Θα ήθελα να καλωσορίσω ορισμένες τροπολογίε για παράδειγμα την νούμερο 2, η οποία αναφέρεται απο... στον αποκλεισμό ε, προσφορών από χώρες της ΕΟΧ και είναι ε, ορθό να μην ακολουθήσουμε τέτοια ε, εκδικητικά ε, μέτρα προστατευτισμού. Χαίρομαι λοιπόν που η συγητής το έχει ξεκαθαρίσει αυτό το σημείο. Πιστεύω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι μπορεί να δημιουργηθεί κίνδυνος για τις επιχειρήσεις ε, εάν υιοθετηθούν τέτοια προστατευτικά μέτρα. Το πρόβλημα που εγώ εντοπίζω είναι η σχέση μεταξύ του άρθρου 6 και του 8 και 10. Φαίνεται ότι ο εισηγητής επιδιώκει να εντείνει αυτήν την ε, σύνδεση και εγώ έχω εκφράσει στο παρελθόν και το επαναλαμβάνω ότι εντιτίθεμαι σε αυτό. Ποιο είναι ο κίνδυνο εάν τα συνδέσουμε αυτά τα άρθρα. Κάποια κράτη-μέλη θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει μια διαδικασία ελέγχου για τις δημόσιες ε, συμβάσεις στη χώρα τους προκειμένου οι αναθέτουσες αρχές στα κράτη-μέλη αυτά να έχουν τη δυνατότητα να αποκλείσουν με βάση το άρθρο 6 προσφορές από τρίτες χώρες. Τώρα η τροπολογία 19 η οποία τροποποιεί το 6 ε, ε, εντείνει αυτή τη, τη, σχέση, γιατί τώρα πλέον θα υπάρχει μια ρητή αναφορά στο άρθρο 8 και αυτό ενθαρρύνει άμεσα τα κράτη-μέλη να ζητούν από την Επιτροπή να ελέγχει τις διαδικασίες στα ίδια. Αυτό ενεντείνει τον κίνδυνο. Αυτό που σας είπε τα κράτη-μέλη δηλαδή να ζητήσουν αυτόν τον έλεγχο προκειμένου να διδώσουν τη δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές τους να αποκλείσουν ορισμένες εταιρείες. Μπορεί να φαίνεται το ζήτημα πολύ τεχνικό, αλλά στην πραγματικότητα θα, δυνατότητα, θα μπορούσε να δώσει δυνατότητα σε ορισμένα κρατημέλη να αυξήσουν τον προστατευτισμό. Τώρα, υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που δεν αναφέρεται σε αυτή την ε, εισήγηση. Θα ήθελα να γνωρίζω εάν θα συζητηθεί φέτος, του χρόνου, οποτεδήποτε, το θέμα αυτό, δεδομένου ότι πολλά κράτη-μέλη αντιτίθενται. Και αναρωτιέμαι επίσης εάν η Επιτροπή έχει αλλάξει την άποψή της δεδομένης της αντίθεσης των κρατών μελών ή αν σκοπεύει να κρατήσει την ίδια θέση επαόριστον. Πιστεύω ότι εμεί θα έπρεπε να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στο άνοιγμα των αγορών μέσω των GPA και όχι σε τέτοια μέτρα προστατευτισμού και καλωσορίζω την έκκληση ο απευθύνει ηγητής να ε, κυρωθεί το, ε, κυρωθούν τέτοιε συμφωνίε, έτσι ώστε να παραμείνουμε ανοιχτοί στο εμπόριο από άλλα μέρη του κόσμου. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, θα συναντηθώ ε, για ένα γεύμα εργασία με την TPC αυτή την εβδομάδα και θα ζητήσω διευκρινήσει σε σχέση με το φακέλο αυτό ο κύριος Ζαντό από τους Πράσινους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στην ε, παρουσίαση του φακέλου βλέπουμε όλες ε, τις δυσκολίες τις οποίες ε, βρισκόμαστε και έχω την εντύπωση ότι αν θα πρέπει να ψηφίσουμε, αν θα πρέπει να ψηφίσουμε εμπιστευτικά, η πλειοψηφία θα πέριπτε την πρόταση της Κομισιόν γιατί δεν απαντά στι προσδοκίες που θα μπορούσαμε να έχουμε και στο τι διακυβεύεται στι προκλήσεις που έχουμε ενώπιόν μα. Μάλιστα, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση και αναφέρθηκε η συνάδελφος από το ΙΣΙΑ στι Συμφωνίες για δημοσιοσυμβάσεις συμβάσει και ταυτόχρονα οι αναδεμινόμενες χώρες είτε βλέπουν τη συμφωνία πολύ μακριά είτε είναι παρατηρητές. Έτσι λοιπόν από τη διεθνή σκοπιά και από τη σκοπιά των ε, αναπτυσσόμενων χωρών αλλά και από τη σκοπιά των βιομηχανοποιημένων χωρών βλέπουμε ότι οι δημόσιες συμβάσεις δεν είναι απλώς ένα επιπλέον εμπορικό εργαλείο όπως σκεφτείτε συχνά η Κομισιόν που πρέπει να το απελευθερώσουμε ε, έναντι ενός δογματισμού ελευθερών συναλλαγών, αλλά ένα εργαλείο βιομηχανικής πολιτικής ε, τη στιγμή που τα κράτη έχουν ε, μικρές δυνατότητες επενδύσεων σήμερα και προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα πολιτικής, δημόσιας πολιτικής που μπορεί να βοηθήσουν στην έξοδο από την κρίση και στην οικοδόμηση μιας αηφόρου οικονομίας. Επομένως, τέθηκαν ε, όλα τα ζητήματα, το θέμα των αναπτυσσόμενων χωρών, των ε, διαδικασιών ε, και των μεθόδων παραγωγής για το τι γίνεται με τις νομοθεσίες σε επίπεδο κρατών μελών ή σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς έχουμε κάποιους δισταγμούς ακόμη από την πλευρά των πρασίνων και δεν θα σας κρύψω ότι είμαστε μεταξύ δύο επιλογών. Είτε ξεκάθαρα να απορρίψουμε την πρόταση της Κομισιόν, εγώ νομίζω στο στάδιο αυτό, γιατί αν λάβουμε υπόψη και την ε, βάση της ε, πρώτης Κομισιόν ε, είναι το να έχουμε ένα άνοιγμα το οποίο θα είναι ούτως ή άλλως καθολικό αλλά θα αποκλείουμε αναπερίπτωση. Όταν ε, σκέφτομαι τη συζήτηση που έγινε στο Συμβούλιο σε σχέση με το πόσο δύναμη είναι η πρόταση Κομισιόν και τη συζήτηση που έχουμε τώρα εδώ μεταξύ μα, ε, το θέμα δεν είναι να καθυστερήσουμε επαόριστον αυτό το ζήτημα, αλλά πρέπει να κάνουμε μια πολύ πιο σοβαρή συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το θέμα των δημοσίων συμβάσεων, ε, για τη χρησιμότητά τους και πώς μπορούν να μας βοηθήσουν οικονομικά πριν απλώς να εφαρμόσουμε το δόγμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή, αλλά και η εισήγηση, η παρουσίαση από την Κρίστα Ρόβολτ δείχνει ότι εδώ έχει γίνει πολύ και ενδελεχής ε, δουλειά και επεξεργασία αυτού του θέματος. Εγώ κοίταξα, ξαναδιάβασα και την εισαγωγή του πρώτου εγγράφου εργασία και τα συμπεράσματα. Και πιστεύω ότι αντανακλά με τον καλύτερο τρόπο ότι ε, την πλεονάζουσα ε, νομοθετική ρύθμιση που υπάρχει, την οποία δεν χρειαζόμαστε, αλλά και στην διαδικασία διαβούλευσης με την Κομισιόν, πάρα πολλές αναθέτουσες αρχές είπαν ότι δεν επισημούν διόλου μία νέα πρόταση και ότι τα πράγματα καλώς έχουν ως έχουν με την παρούσα και ισχύουσα ε, νομοθεσία και τις παρούσες ρυθμίσεις. Γιατί λοιπόν, ποια είναι η προστιθέμενη αξία που προσφέρει τώρα αυτή η πρόταση. Γι' αυτό προτείνω να απορρίψουμε ως Επιτροπή την πρόταση της Κομισιόν, διότι εδώ υπάρχει και ο κίνδυνος μεγάλης ζημίας δεδομένου ότι ορισμένες ε, χώρες αναθέτουσες αρχές μπορούν να, να ερμηνευθούν ότι ακολουθούν μια πάρα πολύ αυταρχική στάση και αρνητική συμπεριφορά. Αυτή η πρόταση υποτίθεται θα βοηθήσει αναπτυσσόμενες χώρες. Όμως πιστεύω ότι θα τις εξαγριώσει περισσότερο, διότι ε, θα τους δώσει το έναυσμα να υιοθετήσουν ε, η παρόμοια νομοθεσία, παρόμοιες ρυθμιστικές, ρυθμιστικούς κανόνες ε, σε εθνικό επίπεδο και έτσι θα δημιουργηθεί μια διαμάχη μεταξύ των χρόνων αυτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένας πόλεμος. Αγαπητοί συνάδελφος, κυρία Ρόβολτ, μου επιτρέπετε να πω ότι ορισμένα κράτη-μέλη και περιφέρειες, ας πούμε η Ιταλία, παραδείγματος χάρη η Ιταλία ή ε, το Βραδεμβούργο στην Γερμανία, ε, χρησιμοποιεί ε, όλες τις δυνατότητες των δημοσίων συμβάσεων που τους επιτρέπει η κοινοτική νομοθεσία και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τώρα, ο εισηγητής θέλει να ε, αφαιρέσει τη δυνατότητα, την ευελιξία χειρισμού των δημοσίων συμβάσεων ε, που παρέχει η νομοθεσία μας και το δικαστήριο και να ακολουθηθεί, να ακολουθηθεί ένας μόνο μοναδικός και ομοιόμορφος τρόπος προσέγγισης. Ενώ εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό είναι σωστό διότι καθιστά το όλο εγχείρημα λιγότερο ευέλικτο και πολύ πιο περιοριστικό. Και ακριβώς την κατεύθυνση που δεν θέλουμε. Ο πρόεδρος. Η Κομισιόν. Ο κύριος Γέσεν και ο κύριος Μίλε από την Κομισιόν παρακαλώ. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε. Ε, το όνομά σα και τα πρακτικά. Τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Καλώ ορίζουμε λοιπόν αυτή την έκθεση από τον εισηγητή. Γιατί περιλαμβάνει διάφορε ενδιαφέρουσε ιδέε. Καλώ ορίζουμε επίση το γεγονό ότι ο στόχο ε, ε, είναι στην ίδια κατεύθυνση με τη γενικότερη φιλοσοφία της πρότασης τη Επιτροπής. Υπάρχουν ορισμένα σημεία στα οποία πρέπει να τα εξετάσουμε περισσότερο, κυρίως ε, το ζήτημα της, σαφής, της σαφούς σύνδεσης μεταξύ του άρθρου 6 και 8, καθώς και ορισμένα άλλα τεχνικά ζητήματα. Όμως πιστεύω ότι αυτή η έκθεση είναι μια καλή βάση εργασίας και με χαρά θα συνεργαστούμε επ' αυτής. Ίσως ο συνάδελφος θέλει να προσθέσει και κάποια άλλα στοιχεία. Ζάνιβ Ο, Μο, από τη Γενική Εμπορίου. Εμείς επίσης καλωσορίζουμε την φιλοσοφία του εισηγητή και το... θα θέλαμε περισσότερο να ασχοληθούμε με το ζήτημα του πώς οι τροπολογίες που προτείνονται θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο κατακαιρματισμού της αγοράς είναι ένα θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε και με τον εισηγήτη και με τους σκιώδεις, κατά πόσον οι τροπολογίες που προτείνονται είναι εφικτές και κατά πόσον θα ενισχύσουν την κοινή αγορά. Από την πλευρά του Συμβουλίου, αν και δεν, φυσικά δεν μπορούμε να μιλήσουμε εξ του, η Επιτροπή έχει ενθαρρύνει την Προεδρία της, τη Λιθουανική να ξαναξεκινήσει τις σχετικές συζητήσεις στο Συμβούλιο. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει εδώ εκπρόσωπος της ε, Προεδρίας. Πάντως η Επιτροπή θα επιθυμούσε να επανεκκινήσει η συζήτηση στο ε, Συμβούλιο και να υπάρξει πρόοδος. Από ό,τι γνωρίζω υπάρχουν κάποιοι από το Συμβούλιο εδώ, όμως δεν συμμετέχουν ε, στη συζήτηση του Κοινοβουλίου. Ας επανέλθουμε στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι για τις παρατηρήσεις σας και τις ε, συζητήσεις που έχουν γίνει τόσο καιρό ήδη για αυτό το θέμα. Εδώ και μήνες, ε, ε, θα έλεγα την αρχή, πίστευα ότι δεν είναι μόνο ένα πολιτικό θέμα, αλλά και θέμα που άπτεται της εθνικότητος, δηλαδή της δαφικής, αν θέλετε, προέλευσης των, προβλημάτων. Ε, είναι τα κράτη, τα, η θέση τους, η προσέγγιση την οποία έχουν και η στάση που τηρούν. Το θέμα είναι ότι η Κομισιόν θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει τη δυνατότητα παρέμβασης βάσει του άρθρου 6. Αυτά και τα άλλα άρθρα πρέπει να συζητηθούν. Μια πολύ σύντομη παρατήρηση. Όταν λέμε αυτή την προθεσμία των πέντε ετών ε, για την εκτελεστική πράξη, αυτό συμφωνεί απόλυτα, συνάδει απόλυτα με τα TDIs και τις συναφείς διατάξεις, η πενταετής διάρκεια. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση εδώ δεν δημιουργούμε ανασφάλεια, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα μέσα σε αυτό το πενταετές χρονικό διάστημα να δούμε εάν ο κανονισμός αυτός έχει λόγο υπάρξεως, αν είναι λογικά τα αποτελέσματα και σωστά ή όχι. Η προθεσμοί για τις ε, τροπολογίες ε, είναι τη Δευτέρα στις 30 ε, αυτού του μήνα μέχρι τις 6 το απόγευμα και θα ψηφίσουμε σε αυτή την επιτροπή στην τακτική μας συνεδρία στο Νοέμβριο. Λοιπόν, περνάμε στις ψηφοφορίες. Ετοιμάστε τις κάρτες σας. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Καθίστε παρακαλώ. Let's vote. First vote. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τις ε, ψηφοφορίες. Πρώτο θέμα, έκθεση κατίνη, ασφάλεια καταναλωτικών προϊόντων. Είναι το σημείο 14 στην ημερήσια διάταξη. 64 τροπολογίες έχουμε να ψηφίσουμε. Η πρώτη είναι τροπολογία 25. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 27, υπάρχει προφορική τροπολογία μου λένε. Δύο μάλλον προφορικές τροπολογίες. Δεν υπάρχει κάποια ένσταση στο να τις ψηφίσουμε μαζί. Επομένως, 27 μαζί με τις προφορικές τροπολογίες υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 28 και 30 είναι ίδιες. Και 29. Μα συγχωρείτε, 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συντονιτές να σηκώνουν πιο ψηλά το χέρι τους γιατί έτσι είναι πολύ πιο εύκολο να, μετράμε τις ψήφους. Παρακαλώ λοιπόν τα μέλη να σηκώνουν όσο δυνατόν πιο ψηλά το χέρι τους. 29 και 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 34. Καταπίπτει. Και φτάνουμε στην 6. τροπολογία 6 και 40 οι οποίε είναι υπέρ κατά Ήταν ίδια με την τροπολογία 40. Τροπολογία 7 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 44 και 45 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 46 με προφορική τροπολογία, αν δεν υπάρχει ένσταση. 46 ως τροποποιήθηκε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 50 υπέρ, κατά, ε, εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος μου φαίνεται πως απορρίπτεται αλλά δεν είμαι σίγουρος ψηφίζουμε για την τροπολογία 60 έναρξη ψηφοφορίας κλίξη και όντως απορρίπτεται τροπολογία 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το ΕΛΚ τι ψήφισε ρωτά ο πρόεδρος. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Τροπολογία 10. Είμαστε τώρα στις ε, τελογικές σκέψεις. 10 υπέρ. Κατά, εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά εγκρίνεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τώρα πηγαίνουμε στην προφορι... στις προφορικές τροπολογίες. Προφορική 4 για την αιτιολογική σκέψη 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρα η τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τελική ψηφοφορία, έναρξη. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 26 υπέρ, 3 κατά χωρίς αποχές. Συγχαρητήρια στον κύριο συνάδελφο, κύριο Μοσκαρτίνη που βρίσκεται στα αριστερά μου. Πάμε στο σημείο 15 της σημερινής της διάταξης. Έκθεση για την εποπτεία της αγοράς προϊόντων. «93 τροπολογίες. Ας αρχίσουμε. Συμβιβαστική 1. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 40 46 καταπίπτει, 48 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 49 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 50 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 51 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 52 υπέρ κατά αποχές δεκτή. «53 υπέρ κατά αποχές δεκτή». 54 υπέρ κατά αποχές δεκτή 55 Ξεχωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά δεκτό, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά δεκτό. 56 υπέρ κατά δεκτή, 57 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή 60 υπέρ κατά αποχές δεκτή 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 61 υπέρ κατά αποχές δεκτή 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 62 με προφορική τροπολογία, δεν υπάρχει αντίρρηση της τροπολογίας, 62, ως τροποποιηθήσα, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 63, α, καταπίπτει. 64 Και αυτή καταπίπτει. 64. Α, όχι, δεν καταπίπτει. 64. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 65. Ξεχωριστή ψηφοφορία του πρώτου μέρους υπέρ κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 66. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή 67 υπέρ κατά αποχές δεκτή απορρίπτεται απορρίπτεται 67 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές δεκτή 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ κατά αποχές δεκτή 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 74 ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή 75 υπέρ κατά αποχές δεκτή 76 υπέρ κατά αποχές δεκτή 77 υπέρ κατά αποχές δεκτή 78 υπέρ κατά αποχές δεκτή 79 υπέρ κατά αποχές δεκτή 80 υπέρ κατά αποχές δεκτή 81 υπέρ κατά αποχές δεκτή 82 υπέρ κατά αποχές δεκτή 83 πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές δεκτό δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτό 84 υπέρ κατά αποχές δεκτή 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή 85 υπέρ κατά αποχές δεκτή 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή 20 υπέρ κατά αποχές 20, 20, σαν ψηφίζουμε την 20, υπέρ, κατά, άποχες, δεκτή. 21, υπέρ, κατά, άποχες, δεκτή. 89, υπέρ, κατά, άποχες, δεκτή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 91 υπέρ κατά αποχές δεκτή 92 υπέρ κατά αποχές δεκτή 93 υπέρ κατά αποχές δεκτή 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή ε, αιτιολογικές σκέψεις ε, συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 24 24 καταπίπτει. 3. 27. 3 υπέρ κατά έγινε δεκτή, 27 ε, υπέρ κατά δεκτή, 28 δεκτή, 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή 37 υπέρ. Α, να ελέγξουμε. Τη 36 παρακαλώ ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται 36. 37. Απορρίπτεται 9. Υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. 33. Υπέρ 38, συγγνώμη, υπέρ κατά αποχές δεκτή, 39, υπέρ κατά αποχές δεκτή, 40 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 42 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 43 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ε, ας ξαναψηφίσουμε τη 43 παρακαλώ, υπέρ κατά αποχές δεκτή. 44 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ε, τελική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 29, καμία ψήφος κατά μία εποχή, συγχαρητήρια στον εισηγητή. Σημείο 17. Συνέκριση του κυρίου Μέρφη. Λοιπόν, επανέλθουμε στο σημείο 16. Μαρία Μπαντία για το ΚΑΡΣ 2020. Υπάρχει μόνο ένα σύμβαση στην τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε για την 9 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 10 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ελέγξουμε τη 19 άρχεται ψηφορία Πέρα. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Για να αλλάξουμε την 20. Βαλέμσκι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε για την 25. Άρχεται η εφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Για την 28, ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Δύο ισοπαλίες. Μάλιστα. είναι, Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30. Όχι. 37. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 39. Υπέρ κατά εποχέ εγκρίνεται 40 υπέρ κατά εποχέ εγκρίνεται 41 τμήματική ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά εποχέ εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά εποχέ απορρίπτεται Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τελική ψηφοφορία, έρχεται ψηφοφορία. «25 υπέρ, μία ψήφος κατά, τέσσερις αποχές, συγχαρητήρια» στη Μαρία Μπαντία. της εισαγωγής ρυζιού στο Μπαγκλαντές. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. Ελέγχουμε για την τροπολογία 8 έναρξη ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. 12 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 κατά τμήματα ψηφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται που λέγει 13 υπέρ και ε, με ενημερώνει λοιπόν ότι δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα. Το δεύτερο τμήμα παραμένει, ρωτά ο πρόεδρο. Ναι. Ε, τροπολογία 13, δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχή το προείπτωτο. Για το αρχικό κείμενο πρώτο τμήμα δεν χρειάζεται ψηφοφορία. Έτσι λοιπόν ψηφίζουμε μόνο για το δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική νούμερο 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ελεκτρονικός έλεγχος για την συμβαστική νούμερο 1, ένα της ψηφορίας. Πέρα ψηφορίας. Ή απορρίφθηκε τελικά. βαθμολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφορία. Ηλεκτρονικά παραλογικό καλό. Άρχεται ψηφορία. με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος, είναι δύο οι ψηφοφορίες. Πρώτα για την πρόταση της Επιτροπής, πρώτη ψηφορία για την πρόταση της Επιτροπής, πέρας ψηφοφορίες Εγκρίνεται. 27 υπέρ, μία κατά, 2 αποχές. Και τώρα η δεύτερη ψηφοφορία έναξη πέρας ψηφοφορίας. Η 29 υπέρ, 1 κατά. Καμία αποχή εγκρίνεται. Τώρα λοιπόν Ο εισηγητής ε, προτείνεται, κύριε Μέρφυ, προτείνεται να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις. κύριε Μέρφυ. Μόνο μετά την ψηφοφορία των τροπολογιών στην Ολομέλεια. Therefore, uh, Επομένως, εάν αποφασίσουμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις μετά από την ψηφοφορία στην Ολομέλεια, τότε θα μπορούσαμε ε, αμέσως αμέσω να υιοθετήσουμε την εντολή, τη διαπραγματευτική εντολή, η οποία θα ήταν τροπολογίες που θα έχουν εγκριθεί από την Ολομέλεια, προφανώς και η διαπραγματευτική ομάδα, ο συνήθως, θα αποτελείται από τον υποφωνόμενο, τον εισηγητή και τον εισηγητή. Υπάρχει κάποια ένσταση σε αυτό. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Γραμματεία ενημερώνει ότι πρέπει να, αυτή η ψηφοφορία πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά. Ε, Ποιο είναι υπέρ λοιπόν αυτή τη πρόταση που σα έκανα για την ε, εντολή διαπραγματεύση, ε, άρχιτη ψηφορία. Πέρα ψηφορία. 27 υπέρ. Μία αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν. Και περνάμε στο σημείο 18 τη σημερινή διάταξη. 18. Ιούλιου Βίνκλερ, δασμολογικές ποσοστώσεις για τον Ίνο. Τροπολογία 1, υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 2, υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. ομόφωνα δεκτή ή το σχέδιο έκθεση. ομοφωνία. Πρέπει να ψηφίσουμε και την το νομοθετικό ψήφισμα. Πάλι άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας, πέρας της ψηφοφορίας. 26 υπέρ, μία ψήφος κατά Να ξαναψηφίσουμε λοιπόν την εντολή διαπραγματεύσεων να ε, ψηφιστεί στο, στην Ολομέλεια. Άρχεται η ψηφοφορία. Α, πρέπει να το διαβάσω. Είναι υποχρεωτικό λέει ο Πρόεδρος. Προτείνουμε να αρχίσουμε τις επιζημωτές του Συμβούλου και την, και την Κομισιόν ε, φτάνοντας ε, μετά την πρώτη ανάγνωση της συμφωνίας να, να υποβάλουμε αναφορά ε, να, να υποβληθεί στην ίντα η έκθεση για ψήφιση στις 17 Σεπτεμβρίου 2013 μαζί με τις αποφάσεις του Omnibus 1 και 2 και αυτό θα αποτελέσει τη βάση του διαπραγματευτικής, διαπραγματευτικής εντολής. Η διαπραγματευτική ομάδα θα είναι ο πρόεδρος, ο εισηγητής και οι ισχυώδεις εισηγητές. Ψηφίζουμε λοιπόν, την απόφαση αυτή. Ε, υπέρ κατά απο, ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία, πέρα της ψηφοφορίας. 26 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά. Άρα λοιπόν εγκρίνεται η απόφαση για ε, την αρχή των διαπραγματεύσεων, για να ξεκινήσει ο διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Ποιο ζήτησε διαδικαστικό, παρακαλώ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, δεν κατάλαβα πολύ καλά την εντολή. Γιατί είπατε ότι θα ήταν το αποτέλεσμα της ψήφου στην Ολομέλεια. Αυτό που διαβάζετε το αποτέλεσμα της ψήφου στην Επιτροπή. Ποια είναι η ακριβής εντολή. Η εντολή θα είναι η έκθεσή μας με τις ε, τροπολογίες στην Ολομέλεια. Στην περίπτωση που εγκριθεί. Εντάξει, κατανοητό. Item 19. Προχωρούμε στο 19. είναι η έκθεση του Νίκολο Ρινάλντι για την άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης, για την άσκηση και επιβολή διεθνών εμπορικών κανόνων. Τροπολογία 7. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 42. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Υπέρ... 1. Ε, ε, ε, δεκτή. 9. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 10. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβιβαστική 2 ήταν, 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 47 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 50 υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή, Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 13 υπέρ. Α, ε, και 53 υπέρ κατά αποχές δεκτές. 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τέσσερα. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 63 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 7. 23 και 68 υπέρ κατά αποχές δεκτές. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές ε, έλεγχος παρακαλώ της 60 της συμβαστικής 8 άρχεται η ψηφοφορία πέρας της 26 υπέρ, μία κατά, δύο αποχές, κάτι δεν πήγε καλά, δεκτή λοιπόν. 26 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 28 ξεχωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 36 ξεχωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό δεύτερο τρίτο όχι το δεύτερο μέρος Τρίτο, τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές. Το τρίτο, τρίτο τμήμα. Δεκτό. 35. Το πρώτο τμήμα καταπίπτει ψηφίζουμε το δεύτερο. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 10. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 38 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 12, συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Και τελική ψηφοφορία. η πρόταση ως τροποποιηθήσα ψηφίσουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας δεκτή 27 υπέρ καμία ψήφος κατά ε, 3 ε, κατά καμία αποχή Ωραία, ψηφίζουμε το νομοθετικό ψήφισμα. Υπέρ, ε, συγγνώμη, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. 27 υπέρ, 3 κατά, καμία αποχή. Εγκρίνεται. Και πάλι, εάν υπάρχει πρόταση για έναρξη διαπραγματεύσεων Νίκολο, Νίκολο Ρινάλντι Ποια, τι προτείνεις Ευχαριστώ τους λέει λέω συγητής, τους και όλους τη Γραμματεία, την Κομισιόν και όλους που συνεργάστηκαν. Το Συμβούλιο θα πρέπει να έχει την εντολή τέλος Οκτωβρίου, στην Ολομέλεια 2 του Οκτωβρίου για να ζητήσουμε την έναρξη του τριμερούς διαλόγου στην, με, στην πρώτη ανάγνωση. Ωραία, ψηφίζουμε την εντολή λοιπόν έναρξη διαβουλεύσεων, λέει ο πρόεδρος, μετά την, ε, το αίτημα του εισηγητή για να ξεκινήσει η, η έναρξη μετά από την ψήφιση των τροπολογιών στην Ολομέλεια. Τη διαπραγματευτική ομάδα θα είναι ε, πρόεδρος, ε, ο εισηγητής και η ε, Κιώδης. Ο Φρανκ Προύστ, Σάμπιν Κούτας, Ζαν Τζάχραντιλ, Γιάννικ Ζαντό και Χέλμουτ Σόλτς. Εντάξει, ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 20 6 υπέρ 0 ε, κατά μία εποχή. Δεν, ε, δεν έχουμε ακόμα καμία περαιτέρω ανακοίνωση. Μόλις έχουμε τίποτα νεότερο θα σας το ανακοινώσουμε, λέει ο Πρόεδρος. Θα κάνει ο Γιώργος. Έτσι δεν είμαστε. Περνάμε στο 20. Διαπραγματεύσει εν ώψη μερού συμφωνία επενδύσεων Κίνα για μια συμφωνία διμερών επενδύσεων. Πριν να περάσουμε στην ψηφοφορία, η κυρία Γκέλλερ από τους Πράσινους με ενημέρωσε ότι η τροπολογία 60 αποσύρεται. Δεν θα την ψηφίσουμε λοιπόν. Προφορική τροπολογία. Υπαριθμόν 6. Έχει τεθεί σε λάθος σημείο και αποσύρεται από τον κατάλογο και θα ψηφίσουμε την 29. Δεν έχουμε λοιπόν προφορική τροπολογία 6. Διαγράφεται. Και θα ψηφίσουμε αντίθετη τροπολογία 29. Αυτή παραμένει. Αυτός είναι ο πολύ σημαντικός φάκελος. Γιατί θα γνωστοποιηθεί στο Συμβούλιο η δική μας άποψη γιατί αναμένεται να θετηθεί εντολή για τις διαπραγματεύσεις ε, αυτών των ε, συμφωνίων επενδύσεων. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 3, υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αποσύρθηκε η προφορική τροπολογία 6. Περνάμε στην 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Υπέρ. Συγγνώμη.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 για τη συμβαστική 7. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4, υπέρ. Κατά. Ψηφίζει Πάντα η φιλελεύθερη. Για την τροπολογία 4 υπέρ. Μετά. Εποχές. Έλεγχος. Για την προφορική τροπολογία 4 αρχή τη ψηφοφορία. Δεν ψήφισε το άλλο. Πέρασε. Εγκρίνεται. 51. Κατά. Αποχέ συγκρίνεται. Να ελέγξουμε την 51. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 52. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, προφορική τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ελέγχουμε την 61 άρχεται η ψηφοφορία η 60 αποσύρθηκε ψηφίζουμε την 61 ψηφίστε παρακαλώ πέρας εγκρίνεται ομόφωνα γιατί κάποιοι νόμιζαν ότι ψηφίζαν την 60. Παραπλανητικό, λοιπόν εκεί. Συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για την 64 αρχική ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 66. Υπέρ. 66. Σας παρακαλώ. Μπάνω την προσοχή σας, παρακαλώ. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 72 ψηφίστε παρακαλώ πέρασε Εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 8, υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 74, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 77, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ελεγχο για την 79. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Και πάλι. Απαραίτητα 81. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 81. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 82 να επαναλάβουμε. Έκανα λάθο. 82 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Να ελέγξουμε τη συμβαστική τροπολογία 9. Παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 89 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 90. Τμήματική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε την προφορική τροπολογία 3, σχόλιο εκτός μικροφώνου. Δεν θα το ψηφίσουμε λοιπόν. Καταπίπτει, επειδή υπάρχει αντίρρηση. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την 91. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε για την 98 ψηφίστε παρακαλώ πέρας και πάλι απορρίπτεται 99 υπέρ κατά αποχές και πάλι δεν είμαι σίγουρος. Για να ελέγξουμε την 99 παρακαλώ, άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία σε 101-102. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος αυτών των τριών τροπολογιών. Άρχεται η ψηφορία. Πέρασε. Για μια ακόμη φορά απορρίπτεται. 103 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται.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 κατά εποχές απορρίπτεται έλεγχος για την 11 άρχεται η ψηφοφορία είναι σημαντική η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 112 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 113 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται.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 κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 2 υπέρ έλεγχος για 17 άρχεται η ψηφοφορία για 17 πέρας εγκρίνεται συμβαστική 2 υπέρ κατά Εποχέ εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1. Υπάρχουν αντιρρήσει, Όχι, α ψηφίσουμε υπέρ. Κατά Εποχέ εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά Εποχέ εγκρίνεται. Προφορική 2. Υπάρχουν αντιρρήσει, Σχόλιο εκτός μικροφώνου. Αντίρρηση μάλλον ξαφνής ομιλητή. Δεν ψηφίζουμε την προφορική 2. 21 υπέρ κατά αποχέ. Απορρίπτεται. 22. Να ελέγξουμε την 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και πάλι. Απορρίπτεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 24, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την 24. μια ακόμη φορά. Απορρίπτεται την ισοπελία. Ψηφίζουμε Θέλει και ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 22 υπέρ, 2 κατά, 6 εποχές. Συγχαρητήρια στον κύριο Σούλτς. Item 21 is... Yes. 21, 21 uh, σχέδιο έκθεση uh, Frank Proust για τις εμπορικέ σχέσεις Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ιβάν. Πρώτα λοιπόν θα ψηφίσουμε για το προφορικό, προφορικό ερώτημα ηλεκτρονικά, άρχιτη ψηφοφορία για την προφορική ερώτηση ηλεκτρονικά. άρχιδη ψηφοφορία. Και μετά θα ψηφίσουμε τις ε, τροπολογίες. Πέρας ψηφοφορίας. 20 υπέρ 9 κατά καμία αποχή. Επομένως, η υποβολή της ε, προφορικής ερώτησης εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε τις τροπολογίες στο ψήφισμα. 24 υπέρ. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική νούμερα 1 υπέρ τι μου ζητάτε να ελέγξω ρωτάει ο πρόεδρος μόνο τα μέλη του Κοινοβουλίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν ένα ηλεκτρονικό έλεγχο, όχι η βοηθή των πολιτικών ομάδων. Συνεχίζουμε λοιπόν. Συμβαστική 1. Υπέρ κατά Αποχές. Σχόλιο εκτός μικροφώνου. Καλά λοιπόν, ας ελέγξουμε το 25, μιας και τώρα το ζήτησε μέλος του Κοινοβουλίου. Ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν για την τροπολογία 25, ε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορίας. 17 υπέρ, 13 κατά. Εγκρίνεται. Λοιπόν, συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, προφορική 5. Υπάρχει αντίρρηση. Όχι. Ε, προφορική τροπολογία νούμερο 5 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική 2. Υπάρχει αντίρρηση. Όχι. Ψηφίζουμε υπέρ για την προφορική 2. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32. 33 με συγχωρείτε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ας ελέγξουμε για την 34 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 25 λέει ο πρόεδρος, 35 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική 1. Α, υπάρχει αντίρρηση όχι. Ψηφίζουμε για την προφορική 1. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 30 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ελέγχουμε την 38 άρχιτη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορία. απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές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 αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές δεν είμαι σίγουρος ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 15 Πέρα Απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική νούμερο 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική δρομολογία 4. Εάν δεν υπάρχει αντίρρηση, ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τρουλή 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 24 ψηφί υπέρ, δύο, κατά, δύο αποχές, εγκρίνεται. Και προχωράμε στο σημείο 22 της συνεργής διάταξης. Προφορικό ερώτημα για την εταιρική ε... ε συμφωνία. Ανατολική εταιρική σχέση. Άρχεται ψηφορία. Πέρασε Πέρας 25 υπέρ, 2 αποχές, καμία ψήφος κατά. Συγχαρητήρια την εισηγήτρια, την κυρία Αντρικέρα. Σημείο 24 της ημερησίας διάταξης αποφασίσαμε χθε ότι θα το συζητήσουμε αργότερα. Σημείο 23 ήταν αυτό, με συγχωρείτε. Λοιπόν, σημείο 24 η της έκθεση του Ιούλιου Winclaff για τις διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ε, με τη Σερβία καθώς και την προσωρινή ε, συμφωνία. Λοιπόν, το ερώτημα είναι αν θέλουμε να ξεκινήσουμε ε, διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Το άντε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω κάτι σε σχέση με τον τελικό, ε, την τελική ψηφοφορία στην Κίνα. Αντί για τρεις ε, αποχές, είχαμε τρεις υπέρ. ε, πατήσαμε λάθος κουμπί. Ωραία λέει ο πρόεδρος. Ήταν ε, για το σημείο 20 τη διαπραγματεύσεις ενώπιση σύμφωνα της Δημερούς Συμφωνίας Επενδύσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας αφού μας ενημέρωσε λοιπόν δημοσίως και άρα επισήμω το Άλντε ότι έγινε λάθος στην ψηφοφορία της ψήφους του, ε, μετράμε, προσμετράμε τις τρεις ψήφους υπέρ και όχι ως αποχές. θα διορθωθεί. Σημείο λοιπόν 24 της ημερησίας διατάξης χρειάζεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για να ξεκινήσει ε, διαπραγμάτευση σε σχέση με τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σερβίας. Η σχετική, το σχετικό ψήφισμα υιοθετήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2012 και αυτό θα είναι η βάση της διαπραγματευτικής εντολής μαζί με τα αποτελέσματα του Omnibus 1 και 2. Η διαπραγματευτική ομάδα συνήθω θα αποτελείται τον πρόεδρο, την εισηγητή και τον σκιώδη. Ε, άρχεται η ψηφορία. Πέρας ψηφορίας. Εγκρίνεται λοιπόν με 27 ψήφους υπέρ και μία κατά χωρίς αποχές. Και τελειώνει η ώρα της ψηφοφορίας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Όποιος θέλει παρακαλώ να αποχωρήσει από την αίθουσα, να αποχωρήσει ησύχως.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 Λοιπόν, καιρό να ξαναρχίσουμε τις εργασίε μας. Το επόμενο θέμα είναι το 25, πάντοτε σημαντικό θέμα, η τροποποίηση της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσει που είναι μια πολυμερή συμφωνία, όπου συμβαλόμενο μέρος είναι η Ένωση μετά από πολλά χρόνια και πολλές διαβουλεύσεις. Παρακαλώ με παρακολουθείτε, ρωτάει ο Πρόεδρος. Έχετε την καλοσύνη να με ακούσετε. Uh, Okay. I'll do. Uh, I'm I'm asked to to communicate that. Μου ζητήθηκε να σας ανακοινώσω. Α, ότι η ομάδα Γκουε καταψήφισε την προφορική ερώτηση για το Βίλνιους. Σας το είπα. Όπως σας ε, έλεγα, προχωρούμε για στο θέμα 25, κρατικές προμήθειες, δημόσιες συμβάσεις και τροποποίηση της συμφωνίας. Αποφασίστηκε λοιπόν να τροποποιηθεί η συμφωνία μεταξύ των συμβαλωμένων μερών και μας ζητήθηκε από την ίντα δηλαδή να στείλουμε την, την ε, άποψή μας στο Συμβούλιο. Είναι πολυμερής αυτή η συμφωνία. Μόνο ε, η, τα, θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνουν μέρος και αυτό άπτεται και της συμφωνίας στο Μπαλί του ΠΟΕ βάσει αυτής, αυτών των συμπερασμάτων αυτής της φωνίας ε, το, ε, ενεργούμε τώρα. Η τροποποίηση τη συμφωνία θα τεθεί ενισχύ αν τα δύο τρίτα των συμβαλλημένων μερών την επικυρώσουν ε, και είμαστε αισιόδοξοι. Είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι θα επιτύχουμε τα δύο τρίτα ο εισηγητής μας. Είναι ο Χέλμουτ Σούλτς, ο οποίος τώρα που θέλω να του δώσω το λόγο, δεν είναι στην αίθουσα. Και ενώ ήταν μέχρι τώρα. Παραμένει όμως η σημασία του θέματος. Δεν νομίζω ότι το Κοινοβούλιο έχει οποιοδήποτε λόγο να απορρίψουμε αυτήν την πρόταση τροποποίησης της συμφωνίας. Ας ακούσουμε λοιπόν την άποψη των πολιτικών ομάδων. Το ΕΛΚ παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εκ μέρους της ομάδας μας μπορώ να πω ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το θέμα αυτό ως έχει. Δεν θέλουμε να παρέμβουμε περαιτέρω. Έχει διαρκέσει εδώ και πολύ καιρό αυτή η διαπραγμάτευση και έχουν επέλθει πολλές βελτιώσεις. Όπως ξέρετε ξεκίνησε με το γύρο της Ουρουγουάης, μετά η τέση ενισχύει τον 96, εν συνεχεία βεβαίως με την πρόοδο των ηλεκτρονικών μέσων, ευρυζωνική, ίντερνετ κλπ. Όλα αυτά εσυ εξελίξεις ενσωματώθηκαν ως βελτιώσεις στη συμφωνία. Υπάρχουν πάρα πολλά συμβαλόμενα μέλη, οι διαβουλεύσεις τράβηξαν πολλά χρόνια και πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε τώρα να καταλήξουμε ε, έχουμε σημειώσει αρκετές επιτυχίες θα έλεγα, σημαντικές επιτυχίες ε, Παραδείγματο χάρη έχουμε διευρύνει την πρόσβαση σε πάρα, ε, σε πάρα φορούς, φορείς. Έχουμε σημειώσει επιτυχίες στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Ε, έχουμε επιβάλει περισσότερη διαφάνεια, μεγαλύτερη διαπραγματευτική ταχύτητα, καλύτερη δωρεάν πρόσβαση και σε δεδομένα και ευκολότερη πρόσβαση και στο κοινό και στους ενδιαφερόμενους φορείς, εταιρείε κλπ. Και είναι πολύ σημαντικό για μας να διευρύνουμε την πρόσβαση στις αγορές που δίνει την ευκαιρία 300, ε, αγορές 300 δισεκατομμυρίων. Οπότε με όλες αυτές τις επιτυχίες που έχουν και την πρόοδο που έχει σημειωθεί δεν νομίζω ότι πρέπει να καθυστερήσουμε άλλο και ε, πιστεύω ότι όλοι είμαστε πεπισμένοι για την αξία αυτής της ε, πρότασης ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και καλό είναι να την υπερψηφίσουμε όσο έχει σήμερα. Α, γύρισε ο εισηγητής μας, ο κύριος Σούλτς και του δίνω το λόγο. Χέλμουτ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε προσπάθησα με αυτήν την πρόταση να προσφέρω ένα συμβιβασμό, μία συμβιβαστική ε, λύση σε όλες αυτές τις διαβουλεύσεις που έχουν γίνει. Όπως ξέρετε και η Κομισιόν, το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη έχουν εκφράσει πολλαπλώς τη διάθεσή τους να καταλήξουν σε μία συμφωνία στην Υπουργική Διάσκεψη αργότερα το Δεκέμβρη στην Ινδονησία και πιστεύω ότι όλοι συμφωνείτε ότι το θέμα αυτό είναι σημαντικό. Ε, αντιμετωπίζουμε πολλές ε, προκλήσεις, ιδίως στις τελωνιακές συμφωνίες με την έκθεση Crossbar, τις οποίες έχουμε συζητήσει. Τώρα λοιπόν έχουμε αυτή την πρόταση τροποποίησης στο τραπέζι που είναι πολύ καλύτερη από αυτή που είχαμε ιδίω όσον αφορά τα πρότυπα, τα, οικο, εκλογικά κριτήρια που έχουν συμπεριληφθεί, τα πρότυπα για τις διασφάλιση της προστασίας εργαζομένων και όλα τα συναφή θέματα. Και γι' αυτό, έχοντα υπόψη αυτή την προσέγγιση, προτείνω να υπερψηφίσουμε την έκθεση, γνωρίζοντας βεβαίως ότι το ποτήρι ακόμα είναι μισογεμάτο. Αλλά αυτή τη στιγμή μπορούμε να, συμβάλλουμε στην βελτίωση δεδομένου ότι οι προτιμησιακές αυτές συμφωνίες μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω τους δεσμούς μας. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Χωσέ Αντρές, η κυρία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όλοι τονίσατε το πόσο σημαντική είναι αυτή η Διεθνής Συμφωνία λόγω των επιπτώσεων που έχει από την οικονομική σκοπιά να διαχειριστεί την οικονομία, να προωθήσει την απασχόληση που είναι θεμελιώδες, ε, τα κράτη ε, υποστηρίζουν ότι θα μπορούσαν οι εξαγωγές να αποτελέσουν μια λύση στην κρίση. Αυξάνεται εδώ η διαφάνεια και ισότιμη μεταχείριση με αυτήν την έκθεση. Υπάρχουν δύο όμως μελιώδη που θέλω να τονίσω. Ένα, ο ρόλος του Κοινοβουλίου πρόκειται εδώ για θέμα γνωμοδότησης, πρέπει να πούμε ναι ή όχι. Η Επιτροπή Ανάπτυξης ζήτησε να έχουμε αυτή την έκθεση. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ψήφισμα, αλλά δεν μπορεί το Κοινοβούλιο να χάσει το ρόλο της παρουσίας και της εποπτείας μιας ε, τέτοιας συμφωνίας με αυτά τα χαρακτηριστικά, καθώς είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή τη στιγμή και λόγω οικονομικής συγκυρίας. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές και εργασιακές πτυχές έχουν βελτιωθεί μεν, αλλά αν εμείς δεν συμμετέχουμε πώς θα γίνει ο έλεγχος. Αυτή είναι μια ερώτηση που τη θέσαμε στην Κομισιόν και θέλουμε να απαντήσουμε και ποιο ρόλο θα παίξουμε εμεί, αν πούμε μόνο ναι ή όχι. Θεωρώ λοιπόν ότι ω κοινοβούλιο, ω θεσμό, ε, δεν μπορούμε να παραιτηθούμε από το να γνωμοδοτήσουμε και αυτό δεν σημαίνει παρέμβαση ούτε καθυστέρηση, αλλά θέλουμε να έχουμε παρουσία και πώς ε, θα ελέγξουμε την υλοποίηση αυτών των συμφωνιών. Αν μπορεί να μας ενημερώσει η Κομισιόν σχετικά. Ευχαριστώ θα ακούσουμε αργότερα την Κομισιόν για το θέμα αυτό. Τώρα, ας ακούσουμε εκπροσώπους των υπόλοιπων πολιτικών ομάδων, το ECR. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ να υποστηρίξω την εισηγητή, να συστήσουμε, να συνενέσει θετικά στην ε, επικύρωση αυτών των συμφωνιών. Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά που έχουν τροποποιηθεί και μπορώ να τα υποστηρίξω. Δηλαδή είναι φανταστικό το ότι μπαίνουν οι αναπτυσσόμενες χώρες, θα τις βοηθήσουν να πτυχθούν οικονομικά, όπως και θα βοηθηθούν όσοι είναι ήδη μέλη για την πρόσβαση σε νέες αγορές. Υπάρχει λοιπόν αμοιβαίο εκεί. Επίσης καλωσορίζω τις ηλεκτρονικές δημοκρασίες και τις νέες βάσεις δεδομένων, γιατί νομίζω ότι θα βοηθήσουν και τις δικές μας επιχειρήσεις να επιταχύνουν τη διαδικασία γιατί μερικές φορές ε, καθυστερούν πάρα πολύ οι διαδικασίες αυτές και οι πρόσθετες υπηρεσίες έχουν προωθηθεί και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι υπάρχει και επέκταση της κάλυψης για τις τηλεπικοινωνίες, γιατί αυτό είναι ένα παράδειγμα ε, ανοίγματο στις δημόσιες συμβάσεις και νομίζω ότι πρέπει να το υποστηρίξουμε. Και Νομίζω ότι πρέπει να κυρώσουμε αυτό το πρωτόκολλο ω Ένωση πριν από τη συνάντηση στον Παλί το Δεκέμβριο και πριν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσει για την πρόσβαση των χωρών ε, σε ό,τι αφορά του ευρωπαϊκού διαγωνισμού. Γιατί, όπω ξέρετε, εγώ είμαι κατά αυτού και πιστεύω ότι αυτή είναι η προτεραιότητα και αυτό είναι ο δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για να δούμε πώ θα τροποποιήσουμε τη Συμφωνία για τι Δημοσίε Συμβάσει και η κυρία Γκοσποντίνοβα είναι εδώ από την Κομισιόν. Καλημέρα σας. Ε, λέγομαι Αριάνο και προέρχομαι από τη Δέλτα Μάρκτ. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Συγητή και τα μέλη αυτής της Επιτροπής ε, για την εξέταση αυτού του φακέλου και επίσης ευχαριστούμε και την κατανόηση της πίεσης που δεχόμαστε από τη Διεθνή Μέρη. Θέλω να απαντήσω στην ερώτηση που τέθηκε και να πω το εξή, η Κομισιόν ε, βεβαίω γνωρίζει πλήρω ότι θέλει να ενημερώνεται το Κοινοβούλιο για την εφαρμογή τη συμφωνία και η Κομισιόν θα εκπροσωπήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Επιτροπή για τη Συμφωνία για τι Δημόσιε Συμβάσει, GPA, και θα ενημερώνει πλήρω ε, το Κοινοβούλιο για την πρόοδο, για το έργο τη Επιτροπή ε, και για τα έγγραφα που θα αποστέλλονται στην Επιτροπή προ συζήτηση το θέμα του κοινωνικού περιβάλλοντος ε, που έθιξαν ορισμένοι βουλευτές είναι ένα από τα θέματα που συμπεριλαμβάνεται στο μελλοντικό πρόγραμμα της Επιτροπής GPA. Θα, ε, θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε πλήρως τα μέλη αυτής της Επιτροπής για την πρόοδο της εφαρμογής. Σας ευχαριστώ. Uh, well, so far we have not been accustomed to being... Και ξέρετε, μέχρι τώρα δεν ήμασταν συνηθισμένοι σε τέτοια ενημέρωση, απλώς είχαμε μια τεχνική ενημέρωση για την τροποποίηση, αλλά για την εφαρμογή. Είναι δέσμευση της Κομισιόν ότι θα υπάρχει αλλαγή από εδώ και πέρα. Συγγνώμη, αυτό που εννοούσα είναι ότι είναι συνήθως πρακτική της Κομισιόν. Όταν ε, στέλνουμε έγραφα στην Επιτροπή GPA, συνηθίζουμε να ενημερώνουμε τα μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Δηλαδή αυτό που εννοούσα είναι ότι είμαστε πλήρως διαφανείς στις εργασίες μας εκεί. Και θα συνεχίσουμε τη συνήθη πρακτική, αυτά που κάνουμε μέχρι τώρα δηλαδή. Χωσέφα, είσαι ικανοποιημένη από την απάντηση της Κομισιόν μια διευκρίνηση αν πρόκειται να μας εκπροσωπήσουν. Εμείς θα μπορούσαμε να θέσουμε ερωτήσεις σε σχέση με την εφαρμογή της συμφωνίας. Μπορούμε να θέσουμε ερωτήσεις στην Κομισιόν για να μας εξηγήσει εδώ πώς εφαρμόζεται η συμφωνία στα πλαίσια αυτής της Επιτροπής. Και μια άλλη ερώτηση που έμεινε κρεμής. Υπάρχει ένας ρόλος παρατηρητών, παραδείγματος χάρη κάποια μικρά κράτη όπως ο Παναμάς τι ρόλο θα διαδραματίσουν. Μας φαίνεται σημαντικό και αυτό για να είναι παρόν το Κοινοβούλιο και όχι να εκπροσωπείται. Βέβαια, μπορείς να θέσεις οποιαδήποτε ερώτηση στην Κομισιόν. Κομισιόν, κάτι άλλο. Έχετε κάποια περαιτέρω απάντηση, αντίδραση στα σχόλια της ε, συναδέλφου. Απλώς θα παραμένω στο άρθρο της συνθήκης και στο γεγονό ότι η Κομισιόν θα συνεχίσει τη σύνηθη πρακτική. Παρατηρητές μπορούν να είναι μόνο μέρη, δηλαδή κράτη-μέλη που θέλουν να είναι μέρη στο μέλλον και μπορούν να έχουν καθεστώς παρατηρητή. Λυπάμαι λοιπόν, φοβάμαι ότι το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να είναι παρατηρητής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπείται από την Κομισιόν εκεί, αλλά το καθεστώς του παρατηρητή μπορούν να το έχουν μόνο τα κράτη που θέλουν να προσχωρήσουν συμφωνία. Ευχαριστώ κύριο Σόλτς. Uh, I think Πιστεύω ότι είμαστε σε ένα κέριο σημείο της συζήτησης και συμφωνώ με, με αυτά τα οποία τόνισε συναδελφός μας. Ε, πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Και γι' αυτό είπα ότι το ποτήρι είναι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Αλλά το ότι το περιεχόμενο, το τι καλύπτει αυτή τη στιγμή η συμφωνία είναι καλύτερο. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε μια επικοδομητική προσέγγιση παρόλα τα προβλήματα που υπάρχουν. Ε, Ίσως ε, λοιπόν μαζί με την Κομισιόν να αντιμετωπίσουμε την περίπτωση να επανέλθει στην Επιτροπή όταν υλοποιήσει, δεν ξέρουμε πώς και πότε θα υλοποιήσει, αλλά έχουμε το δικαίωμα επαναπομπής και γι' αυτό ε, πιστεύω ότι δεν πρέπει να παρεμποδίζουμε την, την επικύρωση, διότι πιστεύω ότι πρέπει να τηρήσουμε πολύ θετική και επικοδομητική στάση για την επικύρωση. Ο πρόεδρος. Ναι, βέβαια, αλλά δεν υλοποιηθεί ε, η συμφωνία, η προτιμησιακή συμφωνία. Δεν μπορείτε να κατηγορήσετε την Επιτροπή αυτό που θέλουμε εμείς είναι να προχωρήσουμε, να δώσουμε το σήμα για την επικύρωση και πρέπει να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να προχωρήσει η τρέχουσα διαδικασία. Έτσι ώστε να δώσουμε την ευκαιρία στην Κομισιόν να γίνει η επικύρωση, να ολοκληρωθεί η διαδικασία επικύρωσης πριν από τη διάσκεψη των Παλί, που έχει πολιτική σημασία λοιπόν, ολοκληρώσαμε τη συζήτηση και η τροπο, προθεσμία τροπολογιών είναι 18 ε, Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα. 14 ε, Οκτωβρίου ψηφοφορία στην Επιτροπή και Ολομέλεια το Νοέμβριο. Το 28, το 26 αναβλήθηκε όπως αποφασίσαμε χτες και έτσι ε, ολοκληρώσαμε τις εργασίες μας. Θα αντιθούμε στις 3 η ώρα. Ευχαριστώ πολύ.